διακοπή σας συνεδρίαση, τα χθεσινά πρακτικά και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί είναι στη διάθεσή σας. Παρατηρήσεις, αν δεν υπάρχουν, εγκρίνονται τα πρακτικά. Και περνούμε στο πρώτο σημείο της απογευματινής μας ημερήσιας διάταξης. Έκθεση Μετσόλα, Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Η κυρία Μετσόλα, η συγκητρια έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανατέθηκε σε μένα η έκθεση αυτή και κανείς ε, δεν φανταζόταν ε, ότι ε, θα καταφέρναμε έξι μήνες μετά την υποβολή της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξουμε την έκθεση αυτή. Χρειάστηκε λοιπόν να καταβάλουμε πολλέ προσπάθειες, χρειάστηκε να αναλύσουμε όλε τι τεχνικέ πτυχέ και λεπτομέρειε τη πρόταση αυτή, χάρη όμω την ιδιαίτερη επικοδομητική συνεργασία που είχαμε του συναδέλφου εδώ στο Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί ενό νέου συστήματο για το οποίο μπορούμε να είμαστε όλοι περήφανοι. Κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων είχαμε κατά νου ότι θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε αυτού οι οποίοι χρειάζονται προστασία, αυστηρή με όσου είναι παράτυποι μετανάστε και ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί και απαιτητικοί με όσους εκμεταλλεύονται τους πιο ευάλωτους ε, ανθρώπους. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε λοιπόν τώρα τη νέα αυτή νομοθεσία και σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς αρχικά καταφέραμε να επερκεράσουμε όλα τα προβλήματα και καταλήξαμε τελικά σε μια νέα πρόταση για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θεσπίσουμε συγκεκριμένο αριθμό συνοριοφυλάκων προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των εξωτερικών μας συνόρων, προκειμένου να μπορούμε να καταπολεμούμε την διεθνή εγκληματικότητα και προκειμένου να μπορούμε να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα όσων χρειάζονται προστασία και προκειμένου να μπορούμε βέβαια να διαχειριζόμαστε και τη μετανάστευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να έρθουν στο ύψο των ευθυνών του. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο το νέο αυτό σύστημα το οποίο προτείνουμε αυτή τη στιγμή θα είναι αποτελεσματικό. Βέβαια, η νομοθεσία αυτή δεν είναι η μοναδική λύση που χρειαζόμαστε στον τομέα τη μετανάστευση είναι καθοριστική όμω σημασία προκειμένου να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την νομοθεσία αυτή με τι υπόλοιπε νομοθεσίε. Αν αντιμετωπίσουμε ανάλογη κρίση με αυτή που είχαμε το 2015, τότε τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, όπω η Μάλτα ή πολλέ άλλε χώρε, θα μπορούν πλέον να έχουν επιπλέον προσωπικό και θα μπορούν πλέον να έχουν την απαραίτητη συνδρομή την οποία χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτέ τι καταστάσει κρίση. Η νομοθεσία λοιπόν αυτή που έτυχε διαπραγματεύσει διαπραγμάτευση τους τελευταίους μήνες δεν αφορά μόνο τα 10.000 αυτά επιπλέον άτομα. Σημαίνει επίση ότι μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματο επιστροφή για όσου είναι παράτυποι μετανάστε. Μα δίδονται με τη νέα αυτή νομοθεσία περισσότερε δυνατότητε να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη, ιδίω όσον αφορά τον εντοπισμό των παράτυπων μεταναστών. Και μπορούμε επίση μέσω τη νέα αυτή πρόταση κανονισμού να μπορούμε να δώσουμε, να χορηγήσουμε πιο εύκολα συνδρομή προ του νόμου μετανάστε και να του δώσουμε και τα απαραίτητα ταξιωτικά έγγραφα. Έχουμε νέε αρμοδιότητες πλέον για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Μπορεί πλέον ο οργανισμό αυτό να προασπίζει και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων θα πρέπει να προστατεύονται. Απότερο στόχο μα είναι να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία, το οποίο να συνάδει με τι βασικέ ευρωπαϊκέ αξίε, οι οποίε για μα είναι πάρα πολύ σημαντικέ ιδίω για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Και αυτό διότι βέβαια γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη θα πρέπει να προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ο Επίτροπο κ. Σαβραμόπουλο έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, στη γλώσσα σας ε, σας ευχαρίστησα. Πώς ήταν η προφορά μου. Θέλει λίγο ακόμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δεν σας κρύβω ότι τα σύνορα και η ακτοφυλακή είναι ένα βασικό βήμα για μια συνολική πολιτική μετανάστευση. Δημιουργήσαμε και εγκαταστήσαμε και ενισχύσαμε σε χρόνο ρεκόρ τον οργανισμό αυτών με κοινέ προσπάθειες. Γνωρίζοντας πολύ καλά τη συνθετότητα των νομοθετικών διαδικασιών συμφωνούμε όλοι ότι πρόκειται περί κατορθώματος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια κυρία Μέτσολα και όλους τους σκιώδεις και τη Ρουμανική Προεδρία που ε, κατέληξαν σε ισορροπημένη συμβιβαστική λύση επί της πρότασης. Η συμφωνία υπογραμμίζει πάλι ότι, και πάλι όταν συνεργαζόμεθα έχουμε καλά αποτελέσματα και δείχνουμε στους πολίτες ότι η Ένωση είναι πρόθυμη και ικανή για δράση. Όταν η, κρίση κορυφώθηκε στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015, η Ευρώπη ε, κατελήφθη εξαπίνης και δεν ήταν έτοιμη. Αντιμετωπεί με εισρωή παράτυπων ε, εισόδων από Ανατολά και Νότο, από τη Μεσόγειο, ε, καταλάβαμε ότι έπρεπε να αναλάβουμε αποφασιστική δράση. Δεν υπήρχε ε, ενιαίος οργανισμός για τα σύνορα, ούτε υπήρχε, υπήρχαν επιχειρησιακές ικανότητες επιτόπου. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου δεν ήταν κατάλληλο για αυτή τη δουλειά. Τα συστήματά μας πληροφόρησης δεν μιλούν, συνομιλούν μεταξύ τους και οι προσπάθειές μας ε, για να εντάξουμε τρίτες χώρες ήταν κατακαιρματισμένες. Αναγκαστήκαμε να λάβουμε άμεσα μέτρα και μακροπρόθεσμα μέτρα και να εργαστούμε παράλληλα σε όλα αυτά τα μέτωπα. Τώρα, τέσσερα χρόνια αργότερα, Όποιος ε, προσπαθήσει να περάσει παράτυπα τα εξωτερικά μας σύνορα εντοπίζεται, ε, λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και εξετάζεται σε βάθος. Σήμερα έχουμε ένα οργανισμό συνοριοφυλακής ακτοφυλακής ολοκληρωμένο, ε, ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, και συστήματα πληροφόρηση που γίνονται διαλειτουργικά όλο και περισσότερο. Με τον νέο κανονισμό που συζητούμε σήμερα θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Ένα στοιχείο κλειδί είναι το μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων ακτοφυλάκων που θα δημιουργηθεί γρήγορα και θα αναπτύξει την πλήρη επιχειρησιακή ε, δυνατότητα των 10.000 ατόμων μέχρι το 2027. Όμως θα μπορούμε να παρακολουθούμε ήδη την 1η Ιανουαρίου του 2021 ε, την ε, αύξηση του προσωπικού. Το άλλο στοιχείο κλειδί που αλλάζει τα πράγματα είναι ότι το μόνιμο προσωπικό του οργανισμού θα έχει εκτελεστικές εξουσίες. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει διαχείριση συνόρων, καθήκοντα επιστροφών, αυτοδικαίως. Βέβαια, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής θα παραμείνουν υπεύθυνες και θα διοικούν και θα ε, είναι επικεφαλής στις δραστηριότητες των οριοφυλάκων και ακτοφυλάκων που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος τους ενώ θα είναι ε, υπό το κράτος μέλος υποδοχής κάποια ε, ε, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνεται έλεγχος σε έγγραφα ταυτοτήτων να υπάρχει άρνηση της εισόδου να σφραγίζονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα να σταματούνται άτομα που παράτυπα επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα και να υπάρχει και ε, υποστήριξη σε διαδικασίες επιστροφών και από άλλες ε, χώρες, από προσωπικό από άλλες χώρες ε, ή για υπηκόους που επιστρέφουν με αναγκαστικά μέτρα. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζονται και θα γίνονται σεβαστά τα ε, υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και θα υπάρχει σωστή ε, κουλτούρα επιχειρήσεων. Ο οργανισμός θα στηρίζει περισσότερο τα κράτη-μέλη στις επιστροφές για να βελτιώνεται η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ε, εμένουσες προκλήσεις μεταναστευτικές. Χαιρετίζω κι άλλες εξελίξεις που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια αυτού του κανονισμού όπως εξυγχρονισμός του παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της επιχειρησιακής δραστηριότητας του οργανισμού. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι στην καρδιά όλων των πρωτοβουλειών της Κομισιόν και αυτής. Όλες οι δραστηριότητες του οργανισμού και των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θεσπίζονται στο χάρτη. Ο οργανισμός θα συνεργαστεί στενά με τον μελλοντικό οργανισμό ασύλου για να έχει πρόσβαση στις διαδικασίες του ασύλου. Ο οργανισμός θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε επίσης ότι εκείνοι που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας θα επιστρέφονται με πλήρη σεβασμό τον, επαναλαμβάνω αυτό, πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι όταν θα συγκροτηθεί το επόμενο κοινοβούλιο, η πρόταση σύσταση ε, του, ε, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασύλου θα εγκριθεί σύντομα. Ελπίζω. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι λυπάμαι διότι η δυνατότητα ε, μηνιαίας διαφορικής πληρωμής στο μόνιμο προσωπικό, η πρόταση αυτή δεν διατηρήθηκε στην τελική συμφωνία. Αυτό είχε στόχο να βελτιώσει την ελκυστικότητα του οργανισμού ως εργοδότη, να διασφαλίσει επίσης μόνιμο προσωπικό που θα προσλαμβάνεται έγκαιρα. Ε, σχετικά με αυτό θα δώσω μια διακήρυξη. Τέλος, πολιτική καθοδήγηση για την ε, ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Αυτό σημαίνει σχεδιασμό ικανοτήτων για τον Οργανισμό Συνορφυλακής και Ακτοφυλακής, ε, αυξημένη συνέπεια με τις υπόλοιπες εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Με αυτό τον καινούριο κανονισμό και ο οργανισμός και τα κράτη-μέλη θα έχουν εργαλεία για να αντιδρούν και να προβλέπουν μελλοντικές κρίσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Τέλος, θα βοηθήσει αυτό στη διατήρηση της, ε, ε, του χώρου Σέγγεν ελεύθερης διακίνησης. Θα βοηθήσει στη διατήρηση του χώρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναμφίβολα η νέα εντολή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλάκων Ακτοφυλάκων είναι σημαντικό βήμα ε, ως ευρωπαϊκή αντίδραση για το μεταναστευτικό. Ε, προβλέπεται αύξηση σε 10.000 άτομα, ε, ε, πλοία, αεροσκάφη. Ε, έτσι θα μπορέσει να είναι πιο λειτουργικός οργανισμός και να σώζει και ζωές. Χρειάζονται πόροι. Γι' αυτό αυτό θα λειτουργήσει μόνο αν ε, συμφωνήσουμε σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο πολιετές και διευρυμένο. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αυστρίας, για παράδειγμα, θα ήθελα να πω ότι όποιος θεωρεί σημαντική τη φύλαξη των συνόρων θα πρέπει να πληρώσει και ε, μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Αυτό είναι κομμάτι μόνο μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση και σίγουρα είναι και ε, μια πολιτική που εκφράζει ε, αλληλεγγύη επίσης ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοέλιο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε, κύριε Βραμόπουλε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έγκριση αυτής της νέας ενισχυμένη τη και είναι ένα ιστορικό βήμα για μια κοινή προστασία των εξωτερικών μας συνόρων. Σχετίζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία ε, στο χώρο Σέγγεν. Μιλάμε για 10.000 ακτοφυλακές που μπορούν να μεταφερθούν ε, στις χώρες όπου είναι πιο ευάλωτα τα σύνορα ή όταν προκύπτει κάτι επίγον. Αυτό δεν πρέπει βεβαίως να οδηγεί στα κράτη-μέλη να μην τηρούν τις ε, ε, υποχρεώσεις τους. Τα, τα, μισά από τα άτομα αυτά, από τους οκτωφύλακες, θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Η Πορτογαλία θα είναι έτοιμη το 2021 να στείλει 110 ε, συνοριοφύλακες. Ε, όμως, παραδείγματος χάρη, κάνουμε κάτι, κάποιες υποσχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις οποίες ενδεχομένω τα κράτη-μέλη δεν μπορέσουν να τηρήσουν στη συνέχεια. Οι... Θα έχουν επίσης έναν ισχυμένο ρόλο ε, για την επιστροφή ανθρώπων που παραμένουν παράνομα στη χώρα μας. Το ένα τρίτο των αποφάσεων όμως εφαρμόζονται, των αποφάσεων, αποφάσεων επιστροφής. Για την Πορτογαλία δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Επίσης ε, υπάρχει το θέμα των δευτερογενών μεταφορών μεταφορών, μετα, μετα ε, βιβάσεων και έχουμε δει ότι τέσσερα κράτη-μέλη χωρίς κανένα απολύτως λόγο κατάργησαν τη Σέγγεν. Ε, και να πω κάτι τελευταίο έκανε για τον εισηγητή που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά ο κύριος Νίντερ Μιούλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια, τη Ρομπέρτα Μέτσολα, για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε, χωρίς την οποία δεν θα είχαμε καταφέρει να εκπονήσουμε αυτή την νομοθετική πρόταση. Να ευχαριστήσω όμως και τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, και όλο το προσωπικό του γραφείου του για την πολύ στεναρή υποστήριξή του. Το 2015 αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των μεταναστών που φτάναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να ενισχύσουμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Κατά συνέπεια, το 2016 είχαμε τη νέα πρόταση για τον Frontex. Η υφιστάμενη πρόταση αποτελεί μια θεωρωμένη πρόταση τη προηγούμενη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω ακούσαμε, αυξάνεται το πεδίο εφαρμογή του οργανισμού πλέον και δίδονται περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι, καθώ επίση και περισσότεροι εμπειρογνώμονε και μεγαλύτερο προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων να διασφαλίσουμε ότι ο Frontex θα εξακολουθήσει να σώζει ζωές όσων διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπολοιπόμεθα από την βασική μας αυτή ανθρωπιστική υποχρέωση. Δεν μπορεί ποτέ κυβερνήσεις, υπουργοί να παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές για εσωτερικούς καθαρά πολιτικούς λόγους. Παράλληλα τώρα η πρόταση αυτή δίνει στον οργανισμό αυτό περισσότερες αρμοδιότητες στην εφαρμογή των επιστροφών, για όσους δηλαδή δεν έχουν καταφέρει να πάρουν άσυλο. Αυτό όμως θα πρέπει να ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να δίδεται καμία νομική δυνατότητα στον οργανισμό να συμμετέχει σε επιστροφές από μία τρίτη χώρα προς μία τέταρτη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση αυτή θα ενισχύει τι υποχρεώσει και τι δεσμεύσει του οργανισμού αυτού όσον αφορά τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Τέλο, είναι λυπηρό το ότι ε, ενώ καταβάλαμε προσπάθειε για να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο από την άλλη δεν κατάφερε να καταλήξει μια συμφωνία όσον αφορά το κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση του συστήματο του Δουβλίνου παρεμποδίστηκε τελικά λόγω καθαρά εσωτερικών πολιτικών λόγων και νομίζω ότι ε, και η έγκριση της προκαταρκτικής συμφωνίας ε, όσον αφορά την υπηρεσία αυτή τελικά δεν ευωδόθηκε λόγω εσωτερικών εθνικών εγωισμών. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από την έκθεση, ένα ευρωπαϊκό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων και αυτό σαφώς θα αποσχολήσει και την επόμενη νομοθετική θητεία. Ο κύριος Βίστησεν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τα εξωτερικά σύνορα ε, έως τώρα, από ό,τι φαίνεται, ποτέ δεν ήταν αντικείμενο ε, πραγματικής ε, προστασίας. Αυτό μας λέτε σήμερα με αυτό το νομοθέτημα. Γι' αυτό το λόγο, 18 χρόνια μετά τη Σέγγεν, ήρθε η ώρα νομίζω να έχουμε μια υπηρεσία συνόρων. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το συμβασμό που προέκυψε από τον Τρίλογο είναι ότι φοβούμαστε ότι είναι πολύ λίγα αυτά που προτείνεται και έρχονται πολύ αργά. Πολλές δικλείδες ασφαλείας ε, δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε την επιστροφή σε τρίτες χώρες. Ε, αυτή τη στιγμή εγκρίνουμε μία λύση η οποία όμως δεν θα ικανοποιήσει κανέναν, ούτε τους πολίτες, ούτε θα είναι πιο ασφαλές το Σέγγεν. Ευχαριστώ κυρία Γκρίσπα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Σεπτέμβριο του 2018 ο πρόεδρος Γιούνκερ παρουσίασε μια νέα μεταρρύθμιση της υπηρεσίας Frontex. Και πριν από δύο χρόνια ε, ήμουν εισηγήτρια και είχα χαιρετήσει ε, την το αποτέλεσμα τη πρώτη αναθεώρηση. Στο όνομα τη ομάδα μου σήμερα κάνω πάλι το ίδιο. Σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, σε ένα χρόνο ρεκόρ. Λυπάμαι βέβαια ε, για κάποια σημεία. Παρ' όλα αυτά είμαι ικανοποιημένη για το πόσο γρήγορα μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την εξέταση του ζητήματο αυτού με μια ισορροπημένη προσέγγιση, αποτελεσματική για την προστασία των συνόρων μα, σεβόμενη τα θεμελιώδη δικαιώματα όπω μα το ζητούσαν οι συμπολίτε μα. Σημειώνω κυρίω και χαίρομαι γι' αυτό ότι γίνεται ένα πραγματικό βήμα προ τα μπρο σε δημοσιονομικό επίπεδο, σε επίπεδο δυνατοτήτων δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, όπω μόλι αναφέρθηκε. Δύο στοιχεία θα ήθελα όμω να τονίσω. Χαίρομαι που λαμβάνουμε γνώση τη δημιουργία μια μόνιμη δύναμη που θα αποτελείται από 10.000 ακτοφύλακε και νοριοφύλακε και όπου τα κράτη-μέλη θα οφείλουν να συνεισφέρουν είναι πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό, πιο συγκεκριμένο από αυτήν, το, αυτό το απόθεμα των 1500 ανθρώπων που είναι διαθέσιμο υποτίθεται, αλλά με ένα σύστημα που δεν λειτουργεί. Είναι λοιπόν ένα χρήσιμο, ένα απαραίτητο βήμα και συγκεκριμένο. Δεύτερον, ε, ω εισηγήτρια στην αναθεώρηση, είχα ζητήσει στο τελικό κείμενο να γίνει μια αναφορά στη δημιουργία ενό κέντρου κατάρτιση Frontex. Διότι αν θέλουμε να ξεπεράσουμε ε, την εθνική ε, προσέγγιση για την προστασία των συνόρων, διότι τα κράτη-μέλη προφανώ και είναι αρμόδια και παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όμω, εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον ευρωπαϊκό χώρο ελεύθερη κυκλοφορία, τη Σέγγεν δηλαδή, εάν θέλουμε να είναι όσο γίνεται λιγότερα τα κενά, πρέπει να είμαστε Ευρωπαίοι. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο ευρωπαϊκό. Και η υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί με τι αρχέ των κρατών μελών. Όχι μόνο να τι υποστηρίζει, να συνεργάζεται μαζί του. Για να μπορεί να γίνει όμως αυτό στην πράξη θα πρέπει να αναπτύξουμε μια, μια πραγματική ευρωπαϊκή κουλτούρα σε επίπεδο κατάρτισης. Αυτό ακριβώς ε, ζητεί το κείμενο και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Ρομπέρτα Μετσόλα, την εισηγήτρια, η οποία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έδειξε μεγάλη ενέργεια, αποφασιστικότητα και χάρη σε αυτήν μπορούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Σε λίγες ώρες ε, η ομάδα μου θα υποστηρίξει στην ψηφοφορία αυτήν τη νέα μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αλμπιόλ Γκούθμαν. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Τελειώνει αυτή η θητεία και, και ουσιαστικά όσοι κυβερνούν την Ευρώπη έχουν εγκαταλείψει οποιαδήποτε ανθρωπιά. Πολιτικές που βασίζονται ουσιαστικά στον θάνατο των ανθρώπων στη θάλασσα, ε, στη σκλαβιά τους, ε, τις, ε, τα βασανιστήρια σε κέντρα κράτηση και τον εκτοπισμό του σε χώρε όπου δεν υπάρχουν καμία εγγύηση ότι θα γίνουν σε αυτά τα δικαιώματά του. Είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν ε, ε, τρόποι εισόδου νόμιμοι και ασφαλεί. Ε, δεν υπάρχουν ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Πλέον δεν επιτρέπουμε καν στι μη οργανώσεις οργανώσει να κάνουν τη δουλειά αυτή, η οποία είναι απαραίτητη. Κάποια στιγμή θα, θα περάσουν από δίκη οι πολιτικοί θύμητος για τις πάνω από 17.000 νεκρούς των τελευταίων 5 ετών στη Μεσόγειο. Οι πολιτικές τους που κλείνουν τα σύνορα και που ε, ουσιαστικά υποχρεώνουν τους μετανάστες να παίξουν τη ζωή τους κοροναγράμματα οδηγούν στο θάνατο 10 ατόμων τη μέρα και ο κανονισμός που ε, ψηφίστε σήμερα ουσιαστικά είναι το απάβγασμα αυτής της απάνθρωπης πολιτικής είναι ένα, ε, μια παραστρατιωτική οργάνωση με 10.000 ανθρώπους με 2 δισεκατομμύρια ευρώ προπολογισμό για να ε, κλειδαμπαρώσουν τα σύνορα, για να εκτοπίσουν τους ανθρώπους, για να κλείσουν τους ανθρώπους σε κέντρα ε, ε κράτησης. Είναι ουσιαστικά το ο στρατιωτικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το όνειρο της ακροδεξιάς που το κάνουν πραγματικότητα φιλελεύθεροι σοσιαλιστές και συντηρητικοί. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία και την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Νομίζω ότι είχαμε πολύ επικοδομητική θέση ως Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στη διάσωση και την έρευνα. Εμείς φροντίσαμε η Frontex να έχει κατάλληλη εντολή έρευνας διάσωσης λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης που βλέπουμε να ε, ε, λαμβάνει η χώρα στη Μεσόγειο. Η πλειοψηφία ετάχθη υπέρ αυτών. Αλλά τα κράτη-μέλη ψήφισαν διαφορετικά. Ε, μπλοκάρισαν τις προσπάθειες της εισηγήτριας να ενισχύσουν τη διάσωση στο κείμενο του νομοθετήματος. Και αυτό είναι πρόβλημα πραγματικό. Η Frontex μπορεί να διασώζει μόνο ανθρώπους στα πλαίσια και στα, μέσα στα όρια της επιχείρησης διάσωσης και ε, είναι πολύ μικρή περιοχή, λίγο έξω από τη Σικελία. Δεν είναι αυτή η περιοχή όπου υπάρχει το πρόβλημα. Και πνίγεται κόσμος στη Μεσόγειο. Τώρα που μιλάμε και παρακολουθούμε, ξέρουμε που είναι. Συ... Οι δεδαγμένες είναι σαφείς. Κανείς δεν πάει όμως να διασώσει αυτούς τους ανθρώπους. Οι ε, κυβερνητικές οργανώσεις ε, ποινικοποιούνται, τους παίρνουν τα πλοία, δεν γίνονται επιχειρήσεις και η ε, ε, έρευνα και διάσωση ε, έγινε στη, κοντά στη Λιβύη, αλλά διασώσεις δεν γίνονται, γιατί τώρα ξέσπασε πόλεμος πάλι εκεί. Έτσι παραβιάζεται η υποχρέωση διάσωσης ε, μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρχει στη Μεσόγειο ε, οργάνωση σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, ε, τα κράτη-μέλη δεν, να, δεν είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε με συντονισμένο τρόπο, αλλιώς θα καταρρεύσουν οι αξίες της Ευρώπης μαζί με τους πνιγμένους. Δέχεστε μπλε κάρτα κυρία Κέλλερ. Όχι. Λυπάμαι, προσπάθησα πάντως. Η κυρία Τζέιμις τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Μικρόφωνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μάταιες προσπάθειες να αντιμετωπίσει μια πολιτική μετανάστευση ε, χωρίς νόημα. 11 ε, δις ευρώ δαπανώνται ε, γι' αυτό. Ο Φραντς Τίμερμανς είπε τον περασμένο μήνα ότι η Ευρώπη δεν βιώνει πια την ε, μεταναστευτική κρίση του 2015 και 2016. Ε, ο Λίβιος Πρωθυπουργό όμως ανακοίνωσε ότι 800.000 τουλάχιστον μετανάστες από τη Λιβύη ε, θα προσπαθήσουν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έχουμε 11 δις, έχουμε 10.000 συνοριοφύλακες και οι διακινητές ανθρώπων δεν έχουν καταθέσει τα όπλα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τα δικά του προβλήματα πέραν της μάχης. Τώρα ε, έχουμε ανοιχτή Ευρώπη μετά την πολιτική Μέρκελ η οποία μας δημιούργησε το πρόβλημα αυτό. Ο κύριος έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι φτάνανε όλο και περισσότερα κύματα μεταναστών και προσφύγων που ουσιαστικά επιβάρυναν πάρα πολύ την Ιταλία αλλά και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνιμο αυτό σώμα των 10.000 ατόμων ουσιαστικά θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις εσωτερικές δυνάμεις των κρατών μελών, καθότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να συνεισφέρουν στη στελέχωση αυτού του μόνιμου σώματος. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να ανακουφίσει οικονομικά τα κράτη-μέλη. Πέρα από όλο αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, τα οποία δεν δίνανται να συνεισφέρουν σε προσωπικό ή χρηματοοικονομικά ακριβώ ακριβώ επειδή υπάρχουν πολλοί ευρωπαϊκοί οικονομικοί περιορισμοί όσον αφορά τον εθνικό μα προπολογισμό. Πώ μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικά. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτό το μόνιμο σώμα δεν θα είναι αρκετά αποτελεσματικό. Ενδεχομένω να ήταν αποτελεσματικό στα χερσαία μόνο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματικό και επιχειρησιακό στα θαλάσσια σύνορα. Σε περιπτώσει όπω αυτέ που αντιμετωπίσουμε στην Ιταλία, που βλέπουμε να φτάνουν εκατοντάδε μετανάστε και πρόσφυγε οι οποίοι διασχίζουν ε, την θάλασσα που μας χωρίζει από χώρες όπως η Λιβύη. Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ανανεωθεί η επιχείρηση Σοφία και να καταφέρουμε τελικά εκ νέου να έχουμε θαλάσσιες αποστολές. Αντίθετα, υπαναχωρούμε, οπισθοδρομούμε με τον νέο αυτό κανονισμό. Νομίζω ότι ε, η εθνική κυριαρχία θα μειωθεί εξαιτία του νέου αυτού οργανισμού. Του τελευταίου μήνε η Ιταλία κατάφερε να μειώσει την έλευση των μεταναστών και κατάφερε σε σχέση με το 2017 να μειώσει την έλευση αυτή κατά 80%. Αυτό όμω δεν έγινε χάρη στη μεταναστευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χάρη στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση τη χώρα μου. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό οργανισμό. Ο κύριο Συναδεινό έχει το λόγο για ένα λεπτό κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό έπειτα από πέντε έτη ενεργής παρουσίας χαίρομαι που η πολιτική της ένωσης προσαρμόζεται και αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και όσα οι πατριωτικές φωνές υπεύθυνα απαρέγκλιτα και πιστά δήλωναν και δηλώνουν για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης για τη διασφάλιση των πολιτών μας και των ζωτικών μας συμφερόντων για την ανάσχεση των λαθρομεταναστευτικών εισρωών απαιτούνται ισχυρά και ασφαλή σύνορα υπό εθνικό έλεγχο και απόλυτη αυτονομία δράσεων από πλευρά των κρατών μελών παρά το όποιο κοινό πεπρωμένο η εθνική κυριαρχία που μοιράζεται δεν ισχυροποιείται και δεν πολλαπλασιάζεται. αντιθέτω ασθενεί και απεμπολείται. τα σύνορα δεν ομοσπονδοποιούνται δεν συνδιαχειρίζονται πολύ απλά καταλύονται. επιπλέον η οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση συνόρων είναι ψευδεπίγραφη. τα σύνορα είναι σύνορα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση ή παραποίηση. η ένωση ενδιαφέρεται βέβαια μόνο για την εξασφάλιση των συμφερόντων τη Γερμανία και των στενών συμμάχων δεν κόπτεται για την προστασία συνόρων αλλά για να παρκάρει τους λαθρομετανάστες στις χώρες της περιφέρειας όπως είναι η ελλάδα και η ιταλία. ευχαριστώ. Λένερς, ε, λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα εξωτερικά σύνορα της Ολλανδίας ε, έχουν πάει στη Λαμπεντούζα πια. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και αυτή την πρόκληση θα την αντιμετωπίσουμε μόνο με τη συνεργασία. Αν στο μέλλον θέλουμε να έχουμε όφελος από το Σέγγεν και να μην έχουμε εσωτερικά σύνορα, όταν θέλουμε να ξέρουμε ποιο έρχεται στην Ευρώπη και γιατί, αν θέλουμε να ελέγξουμε τη μετανάστευση και να διασφαλίσουμε ότι όσοι δεν έχουν άσυλο θα επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης, αν τα θέλουμε όλα αυτά, τότε είναι σημαντική η ενίσχυση του Οργανισμού Συνοριοφυλακής Ακτοφυλακής. Αυτοί οι 10.000 χρειάζεται να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα και αυτός είναι και τρόπος οργάνωσης της διαχείρισης των σύνορων μας. Διότι είναι καλό να υπάρχει κάτι όχι ε, μόνο όταν χρειάζεται, αλλά να υπάρχει μια μόνιμη βάση υποστήριξης. Το μόνιμο σώμα θα βοηθήσει εδώ. Θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες η ακτοφυλακή και η συνοριοφυλακή να συνεργάζεται με τρίτες χώρες και να τις βοηθάει τις τρίτες αυτές χώρες για να σταματάει η παράτυπη μετανάστευση και να διασφαλίζεται η επιστροφή των ανθρώπων αυτών. Είναι σημαντικό και αναγκαίο βήμα αυτό για την βελτιωμένη επιτήρηση των συνόρων. Να βελτιώσουμε τη διαχείριση των συνόρων. Ευχαριστώ τη Ρομπέρτα Μέτσολα για ε, ε, την ε, αποτελεσματική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική ενίσχυση του Οργανισμού Συνοριοφυλακής Ακτοφυλακής. Ορισμένα κράτη-μέλη όμως μπερδεύουν τα ασφαλή σύνορα με την πλήρη απομόνωση και ε, έτσι καταδιώκουν ανθρώπους ε, και τους στέλνουν στα χέρια των διακινητών. Η, τα, η, απόρρια αυτής της πολιτικής φαίνεται στη Λιβύη τώρα. Δεν φτάνει ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν αναλαμβάνουν τις χριστιανικές τους ε, ευθύνες, αλλά αν ε, ακολουθούσαμε τους ε, συντηρητικούς θα έπρεπε να αναθέσουν τις επιστροφές σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μεταθέτει δηλαδή ίδιες ευθύνες σε άλλους. Αυτό το απορρίψαμε με επιτυχία. Το Συμβούλιο που λάμπει σήμερα δια της απουσίας του πότε θα ε, ολοκληρώσει ένα πακέτο για το ε, άσυλο που θα είναι ισορροπημένο. Πότε θα υπάρξουν ενιαίοι κανόνες για την νόμιμη μετανάστευση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο βιώσιμο και μακροπρόθεσμο τις προκλήσεις στα σύνορα και θα ε, ανταποκριθούμε και όπως πρέπει στις κοινέ μας αξίες. Δέχεστε μπλε κάρτα από την κυρία Σόιντροβα. Οπωσδήποτε όχι, ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ε, Μπέρντ Κέλμελε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση η Frontex και προσωπικό περισσότερο χρειάζεται. Είναι σωστό το μέτρο. Παράλληλα ε, οι 10.000 ε, δημιουργούν ένα πρόβλημα. Τα προβλήματα της Ένωσης δεν θα τα λύσουμε ε, ζητώντας μόνο περισσότερα χρήματα. Αυτό που χρειάζεται για τη μετανάστευση είναι μία ρύθμιση νομοθετική ευρεία που θα δώσει τη δυνατότητα ανάληψης δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.